κύριε Η συζήτηση λοιπόν για την Αίγυπτο έχει τελειώσει. Η επόμενη συνεδρία σε ολομέλειες είναι αύριο από τις 9 έως τις 2 και από τις 13 μέχρι τις 19 έχει εξαντληθεί η ημερήσια διάταξη και θα είναι η ημερήσια διάταξη θα είναι